εμείς τις τελευταίες εβδομάδες και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Ας προχωρήσουμε λοιπόν και ας δράσουμε. Ευχαριστώ ε, κυρία Ρέντινγκ. Η συζήτηση τελείωσε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους και την επιμελητία και διερμηνία για την υπομονή τους.